So, uh, Καλημέρα σας, συνάδελφοι. Έχουμε σήμερα κοινή συνεδρίαση το πρωί για τους κοινούς φακέλους με την ΔΕΒΕ. Έχουμε διερμηνία σε 21 γλώσσες. Τα έγγραφα της συνεδρίασης είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και η συνεδρία θα καλύπτεται μέσω web streaming σωρίζω άπαντες. Ελπίζω να έχετε έτοιμες τις κάρτες ηλεκτρονικής σας ψηφοφορίας. Ξεκινώ με την τροπολογία 91, υπέρ. Κατά. Αποχές. Α. Να την ελέγξουμε. It happens sometimes. So, the Πέρας. Ποιος μιλάει εκεί πίσω. Κυρία Μάης να ψηφίσετε υπέρ ή κατά. Εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. It's closed. Πέρας. <clears throat> Εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά Αμαχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, Αμαχέ εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 113 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε, να επαληθεύσουμε παρακαλώ. And it's closed. Πέρασε. Εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 141 τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. The vote is closed. Πέρας. Εγκρίνεται. 141 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 142 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές να επαληθεύσουμε την 146 παρακαλώ. Καλημέρα σας κυρία Γιώσο. Πέρασε. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. Σημαστική 12 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 165 ε, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κα... υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε. Πέρας εγκρίνεται 168 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ. Κατά αποχές να επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 όχι καταπίπτει. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 σε δύο τμήματα. Πρώτο με προφορική τροπολογία που την έχετε στον κατάλογό σας έχει κάποιο αντίρρηση προς την προφορική. Επομένως, μαζί με την προφορική υπέρ. Πρώτο τμήμα, μαζί με την προφορική υπέρ. Ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Κάτι λέγεται εκτός μικροφώνου. Πρόκειται για ψηφοφορία κατά τμήματα. Στο πρώτο τμήμα έχουμε προφορική τροπολογία. Εφόσον δεν έχουμε αντίρρηση, Ψηφίζουμε μαζί με την προφορική τροπολογία το πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε παρακαλώ το δεύτερο τμήμα. Απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 205 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 216 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.18 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.19 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.21 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.24 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πού βρίσκομαι. Α, 2.30. 2.30 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Θέλετε τη 2.29 να ελέγξουμε. Παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.39 πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.41 υπέρ κατά να ελέγξουμε παρακαλώ πέρασε εγκρίνεται συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.48 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.58 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε την 2.58. Πέρας, εγκρίνεται. 2.60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.63 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.56 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.59 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.64 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 275 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 276 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 277 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 278 εγκρίνεται και περνάω τώρα στην πρόεδρο της ΔΕΒΕ για την υπόλοιπη ψηφοφορία Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 καταπίπτει και περνάμε στην 3, 2 και 7 είναι ταυτόσιμε. Υπέρ, κατά, απόχέ εγκρίνονται. 19. Υπέρ, κατά, Αποχέ, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 11 και 12. Υπέρ, κατά, άποχέ, εγκρίνονται. 13. Υπέρ, κατά, απόχέ. εγκρίνεται νομίζω, αλλά ελέγχουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 22 άρχιδη ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 23. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 54 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα της 54. Πέρες ψηφοφορίας. 55. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Αν δείχνετε τι ψηφίζετε θα με βοηθούσατε. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Στην 66. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Πρώτο τμήμα της 66. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνατε. 30 με 29 κατά. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65, υπέρ. Κατά. Αποχές, επαλήθευση 65, άρχιτη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. 70. Υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ψηφίζουμε την 70 πέρας απορρίπτεται Συμβιβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε είναι 75. Πέρας. Εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίσουμε την 81. Πέρας απορρίπτεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τελευταία σελίδα 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Ε, εγκρίνεται. 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Νομίζω με ίδια πλειοψηφία θα εγκριθεί. Πέρας. Όχι, απορρίπτεται. Μάλιστα. Τελική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεσης όπως έχει τροποποιηθεί με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε με 57 ψήφους υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια στους εισηγητές. Yeah, thank you to the... Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Περιβάλλοντος για τη συνεργασία σας. Είναι η τελευταία φορά που συνεδριάζουμε από κοινού. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ συνάδελφοι. Και εμείς έχουμε ψηφοφορίες, όμως στις 10. Αν θέλετε μπορούμε να ψηφίσουμε αμέσω. Δεν επιτρέπεται αυτό. Αν οι πολιτικές ομάδες θέλουν να παραμείνουν και να ψηφίσουν για την Επιτροπή Περιβάλλοντος, τώρα, όχι στις 10, μπορούμε. Ωραία λοιπόν, θα δώσουμε δύο λεπτά χρόνο στους συναδέλφους της Επιτροπής Ανάπτυξης να αποχωρήσουν από την αίθουσα και μετά ψηφίζουμε. Um, okay, so uh, the good news is we have only two... Μάλιστα, έχω καλά νέα. Μόνο δύο ψηφοφορίες έχουμε για σήμερα, οι οποίες όμως θα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά. Uh, madam. I have uh, still? Thank you. I was. We have to change the machine. Πρέπει μάλλον να αλλάξουμε τα μηχανήματα έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν διαφορετική σύνθεση ψηφοφορίας.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 So I'm asking you again, are there objections to take the vote? Συνάδελφοι, υπάρχουν ενστάσεις ε, για να γίνει η ψηφοφορία τώρα. Οι πολιτικές ομάδες, τι λέτε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από ό,τι μου λένε, αλλά όπως θέλετε θα κάνουμε. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία, η πλειοψηφία των πολιτικών ομάδων συμφωνούν να γίνει τώρα η ψηφοφορία. Η πρώτη λοιπόν That's because we don't have uh, policy advisors. Ε, ναι, δεν υπάρχουν οι σύμβουλοι πολιτικής, δεν παρίστανται. <coughs> Yes, but we have uh, the shadow rapporteur for the first one. Είναι εδώ ο σκιώδης εισηγητής για την ε, πρώτη έκθεση. Hey, so look at the shadow rapporteur, huh? or uh, the coordinator, depending who's present. Ωραία, λοιπόν, οι σκιώδεις εισηγητές, οι συντονιστές, ποιος είναι παρόν. Κυρία Ντάλη, συμφωνείτε με τη διαδικασία, θέλετε να ψηφίσουμε. Ωραία, Ψηφίζουμε, λοιπόν για την ε, προσωρινή συμφωνία για τις ε, διοργανικέ διαπραγματεύσεις για τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα των νέων βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Okay, the vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερη ψηφοφορία πάλι για την προσωρινή συμφωνία που προέκυψε από τις διοργανικές διαπραγματεύσεις, αυτή τη φορά για την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνατε. Και αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε στις 10 για την ανταλλαγή απόψεων με το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο όσον αφορά το ενωσιακό σύστημα μέτρησης εκπομπών ρήπων των οχημάτων.